Dear colleague, please, we have to... Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αρχίσουμε με τις... Per favore, potete... Nell'apposita Σας παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική σας κάρτα. Nell'apposita fessura. Fessura. Se ho la vostra attenzione. Λοιπόν, θα ήθελα να αρχίσουμε με τις ψηφοφορίες. Σας παρακαλώ πολύ ως προς την έκθεση για τη σύσταση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας. Ο Σερ Γκρέιαμ Βότσον είναι μαζί μας και μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία σας, Σερ Γκρέιαμ. Μπορούμε να αρχίσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία αυτή. Αρχίζουμε με την τροπολογία 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 27 η οποία είναι και προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 ε, ε, όχι, όχι, περνάμε στην 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε την 33. Αρχίζει η ψηφοφορία. 49 ε. Κλείνει η ψηφοφορία 34 υπέρ 15 κατά 34 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι εγκρίνεται θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά πολύ ευχαρίστως για την 34 αρχίζει η ψηφοφορία Ας ελέγξουμε. Beh, manca ancora uno, comunque chiudiamo la votazione. Λείπει ένας, αλλά κλείνουμε. Ecco, adesso sono 52-52. Chiudiamo, sì, chiudiamo. Πέρας. Εγκρίνεται 28 υπέρ, 24 κατά. Συμβιβασμός 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44. Τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε την 37, την οποία ξεχάσαμε. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47. 46 θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία και αρχίζει. Non la 28 υπέρ, κατά 26, δύο αποχές εγκρίνεται. 47. Όχι, κάνω λάθος. 49, 49. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 2, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 52, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές δεν είμαι απολύτως σίγουρος, άρα ελέγχουμε ηλεκτρονικά. La votazione. 32 υπέρ, 29 κατά, εγκρίνεται. Άλλη μια ψήφος που πρέπει να προσθέσω. Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Άρα επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία για την 79 ηλεκτρονικά. Ωραία. Εντάξει. εγκρίνεται 32 υπέρ κατά 27. Αποσύρεται 80-81 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 85 κατά πίπτη 86 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές μου φαίνεται ότι έχει εγκριθεί. Δεν συμφωνείτε. Καλά. Ας ελέγξουμε λοιπόν. 87 αρχίζει η ψηφοφορία. Έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Ψηφίζουμε. 87. Πέρας. Απορρίπτεται με 39 ψήφους κατά 21 υπέρ. 89 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 90-91 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19. Μα είχε εγκριθεί το 18. Μπας περιπτώσει, ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 18 ψηφίζουμε. Chiusa la votazione. Πέρας. 32 υπέρ, 28 κατά. Όχι με μεγάλη διαφορά. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 13. 13. Πέρας. 31 έναντι 26 εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θα σας πρότεινα να ψηφίσουμε unblock, αλλά η απάντηση είναι όχι. Εγώ κατάλαβα ότι όχι. Ωραία. Μπορούμε να ψηφίσουμε unblock. Ένα με έξι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. ναι, έχετε διέστηση βλέπω. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική, η οποία και αρχίζει. Διαβάζετε τη σκέψη μου. Ωραία. Ε, σερ, σερ και το αξίζει. 54 ψήφοι υπέρ, ένας κατά. Πάρτε και την ηλεκτρονική σας κάρτα, μην την ξεχάσετε και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τις εργασίες μας λοιπόν. Αρχίζει η συζήτηση για την Περιφερειακή Σύμβαση για τους προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής σε πανευρο... βάση. Όποιος έχει ακουστικά ακούει. Κολέγα είναι e, eh, Πρόκειται για την ε, πρόταση του Συμβουλίου για την Περιφερειακή Σύμβαση σας παρακαλώ συνάδελφοι. Αποχωρήσατε ησύχω. Πρόκειται για μια συνενετική διαδικασία που αφορά την ΙΝΤΑ, την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Εμείς απλώς γνωμοδοτούμε. Έχουμε το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση της ΙΝΤΑ που ξέρουμε ότι τροποποιήθηκε και ο εισηγητής ζήτησε τη γνώμη της νομικής της νομικής υπηρεσίας, άρα θα γίνει μία μικρή τροποποίηση. Θα γίνει η συζήτηση σήμερα, αλλά ε, ως προς την προθεσμία για τις τροπολογίες θα παραταθεί η προθεσμία. Δεν ξέρουμε όμως μέχρι πότε. Ο κύριος Πεγιόν έχει το λόγο και ελπίζω να τον παρακολουθήσετε με προσοχή. Έχετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, εμείς θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε για μια περιφερειακή ε, σύμβαση για ένα καθεστώς προτιμησιακής ε, ε, αντιμετώπισης είναι τεχνικής φύσεως, πανευρομεσογειακό λέγεται, ε, αλλά όσο τεχνικό και να είναι θα έχει μεγάλη επιπτώσεις, ιδιαίτερα για τις χώρες του Νότου. Η σύμβαση αυτή, για να προσπαθήσω να σας την παρουσιάσω, έχει να κάνει με τους ε, κανόνες προέλευσης. Τι σημαίνει αυτό, να ορίσουμε ποια είναι η χώρα προέλευσης ε, ενός προϊόντος και ε, να είναι και σωρευτική αυτή η διαδικασία γιατί δεν αφορά μία χώρα και μόνο. Σόρευση κανόνων καταγωγής προέλευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχουν οι χώρες που είναι στη διαδικασία της Βαρκελόνης η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ευθέρων Συναλλαγών Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Λιχτεστάιν, η νήσι Φερόε και αυτό είναι η καινοτομία, οι χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, δηλαδή οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Οι στόχοι της σύμβασης, γιατί δεν είναι πάντα γνωστό το αντικείμενο, είναι ο εξορθολογισμός κυρίως, γιατί σήμερα έχουμε πάνω από 100 διμερή ε, κείμενα σε θέματα κανόνων προέλευσης. Ε, και φιλοδοξεί ένα κείμενο να αντικαταστήσει ε, όλα αυτά τα 100 και πλέον. Επίση, ε, ταυτόχρονα θα γίνει μια αναθεώρηση και μια ενημέρωση, μια απλούστευση. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με την προσπάθεια αυτή. Θα επιτρέψει επίση την καλύτερη πρόσβαση νέων εταίρων, όπω είναι η Ουκρανία και α ελπίσουμε κάποια των ημερών και η Λιβύη. και τα Δυτικά Βαλκάνια. Μέχρι τώρα είχαν ε, διαφορετικής φύσεως ε, συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εμπορικές προτιμήσεις. Και τρίτος στόχος είναι η διευκόλυνση των συναλλαγών μεταξύ των χωρών μελών, γνωρίζοντας ότι οι δυνατότητες που προσφέρονται σε κάποιες χώρες του Νότου ε, για να έχουν το προσημισιακό καθεστώς, λόγω του συστήματος γενικά χρησιμοποιούνται λίγο γιατί είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα και δεν χρησιμοποιούν την ατέλεια που έχουν ε, ε, στα τελωνία. Η γνωμοδότηση λοιπόν είναι πολύ θετική και επιθυμώ να την εγκρίνετε διότι οι στόχοι που σας ανέφερα είναι όλοι αξιέπαινοι και πάντα στο βαθμό που συμμετέχουν στην οικονομική ολοκλήρωση της ευρωμεσογειακής ε, ζώνης και είναι από τους βασικούς στόχους ε, της ευρωμεσογειακής πολιτικής μας. Τη σύμβαση αυτή την επιθυμούν και οι χώρες του Νότου και οι χώρες της Ανατολής Ευρώπης εδώ και καιρό και ε, μετά από τις επαναστάσεις στον αραβικό κόσμο ακολούθησαν εξελίξεις που δικαιολογούν την προσπάθεια αυτή και θα ζητήσω σύντομα να εγκριθεί η σύμβαση αυτή με τη δική μας νομοδότηση και την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου. Το πλαίσιο είναι διάζων βέβαια. Όσο θετική και να είναι αυτή η σύμβαση, δεν αρκεί από μόνη της η έγκριση για να ε, γίνουν οι αλλαγές που θα επιθυμούσαμε. Χρειάζεται να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα. Δηλαδή, η σύμβαση για να είναι πλήρη στην ισχύ της ε, έχει κάποιους όρους και προϋποθέσεις και κάποια εμπόδια που πρέπει να αρθούν. Έτσι λοιπόν θα πρέπει και οι χώρες του Νότου της Μεσογείου να ε, άρουν τα εμπόδια μεταξύ τους <laughs> και να υπογράφουν ε, ε, συμφωνίες συναλλαγών με χώρες του Νότου μεταξύ τους. Ξέρετε τι δυσκολίες έχουν οι χώρες του Μαγκρέμπ. Η σύμβαση βασίζεται στην καλή τελωνιακή συνεργασία, ικανοποιητική εφαρμογή των ισχυρών διατάξεων και γέννη στην εμπιστοσύνη μεταξύ των ενεχομένων μερών. Η κοινωνία των πολιτών και οι ενδιαφερόμενοι απευθύνθηκαν επανειλημμένα σε εμά. Ε, ε, κάναμε μια έρευνα στις τελωνιακές υπηρεσίες και είδαμε ότι ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίστηκε το θέμα των εισαγωγών κάποιων προϊόντων ε, από ε, της, ε, τους Ισραηλινούς επικισμούς στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Βέβαια αυτό το κείμενο δεν φιλοδοξεί να λύσει έτσι πολύ βαριά προβλήματα, ούτε να ε, μπούμε σε μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Ζητήσαμε όμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια αντικειμενική όσο και σε βάθος μελέτη για την πραγματική κατάσταση. Γιατί κάπως έτσι δηλητηριάζεται το κλίμα και η έγκριση της σύμβασης αυτής Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη σύντομη κατά τα άλλα παρέμβασή μου, λέγοντας ότι η σύναψη της συμφωνίας αυτής ε, μπορεί να είναι ε, χρήσιμη, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να ακολουθηθεί από κανόνες ε, προέλευση πανευρωμεσογειακή, γιατί οι περισσότεροι κανόνε που έχουμε ανάγονται στη δεκαετία του 1970. Αυτό ο εξυγχρονισμό για μα λοιπόν θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια πιο φιλόδοξη μεταξέλιξη τη εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στου εταίρου τη Μεσογείου και το νέο πολιτικό πλαίσιο καθιστά αυτή την ανάγκη ακόμα πιο επιτακτική. Τέλος, στο μέλλον θα χρειαστεί να αποφαθούμε για το θέμα αυτό πάλι με γνωμοδότηση προσεχώς για την ε, ε, μεσογειακή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη για να μπορεί να είναι στο ύψος των όσων απαιτούνται για να ολοκληρωθούν περισσότερο οι εμπορικές μας σχέσεις με τους εταίρους μας στην Νότια Μεσογείο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ανδρικέν. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκ μέρους της ομάδας του ΕΛΚ είμαι ισχυώδης εισηγητρία για αυτό το θέμα. Κατά την άποψή μου, η ιδέα να διαθέτουμε μία ενιαία σύμβαση για τους κανόνες καταγωγής ε, στην, περιοχή, στην ευρωμεσογειακή περιοχή είναι πολύ καλή. Αυτή τη στιγμή έχουμε 60 διαφορετικές συμφωνίες αυτό δημιουργεί σημαντικά τεχνικά και διοικητικά προβλήματα στους τελωνιακούς υπαλλήλους και στους εξαγωγείς που ε, χάνουν, τα χάνουν μπροστά σε, τότια, σε τόσες συμφωνίες. Η σύμβαση, όπως ανέφερε ο εισηγητής, ε, εντάσσει όλα τα πρωτόκολλα που ισχύουν αυτή τη στιγμή περί κανόνων καταγωγής με όλα τα ενδιαφέρομενα μέρη. Μέσα σε ένα σύστημα, λοιπόν, ενιαίο σύστημα κανόνων καταγωγής για όλη αυτή την γεωγραφική περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο ε, κείμενο, ένα ενιαίο μέσο, ε, μέσω μιας περιφερειακής ε, σύμβασης που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις κατά περίπτωση ζώνες ελεύθερων συναλλαγών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεδομένων των ιστορικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην Ευρωμεσογειακή ζώνη. Το εργαλείο αυτό ε, ενοποίησης ε, θα είναι πολύ σημαντικό για την ε, προώθηση μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών σε αυτήν την περιοχή που είναι ο τελικός μας στόχος. Η ολοκλήρωση όμως σε μια τέτοιου ζώ, ελεύθερη ζώνη δεν μπορεί να γίνει χωρίς κοινού κοινούς κανόνες καταγωγής. Οι Υπουργοί Εμπορίου ήδη στις 9 Δεκεμβρίου 2009 στις Βρυξέλλες υιοθέτησαν, ενέκριναν πολιτικά αυτή την σύμβαση και τώρα ήρθε και η δική μας ε, σειρά. Να σχολιάσω και το εξή, το οποίο κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Διεθνή Επιτροπή Εμπορίου χτες στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου χτες. Ε, η κυρία Κοπά μίλησε εκ μέρους του εισηγητή για αυτό το θέμα στην ΙΝΤΑ ε, εκ μέρους δηλαδή του κυρίου Ντελβάγε μας είπε ότι οι συνάλφοι από τη σοσιαλιστική ομάδα έχουν, έρθει με την, ε, έχουν σε επαφή με την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου προκειμένου αυτή να δώσει την άποψή της για τα προϊόντα που προέρχονται από τους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Προφανώς είναι δικαίωμά αλλά όπως είπαμε και χτες στην Ίντα και όπως επιβεβαιώθηκε και από τον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει συμφωνία με το Ισραήλ που ακριβώς ρυθμίζει το θέμα αυτό. Η συμφωνία αυτή υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ το 2004 και αναφέρει ρητά ότι τα τελωνιακά έγγραφα ε, του Ισραήλ θα περιλαμβάνουν την περιοχή, τη ζώνη ή την πόλη στην οποία έχει γίνει παραγωγή. Και τα, όλα τα, και τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από περιοχές που έχει καταλάβει το 1967 το Ισραήλ δεν θα λαμβάνουν προτιμήσεις, δεν έχουν προτιμησιακή μεταχείριση. Ε, με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η καταγωγή ε, των ε, προϊόντων από αυτές τις ε, ζώνες. Πραγματικά ελπίζω ότι η γνώμη της νομικής υπηρεσία του Κοινοβουλίου δεν θα αργήσει πολύ και δεν θα δημιουργήσει εμπόδια στην υιοθέτηση αυτής της σύμβασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρακτικό αποτέλεσμα της εφαρμογής της σύμβασης θα είναι μια ισχυρή όθηση στο εμπόριο και τις ανταλλαγές, καθώς επίσης και σε πιο ισχυρές πολιτικές σχέσεις. Τέλος, να πω ότι είμαι υπέρ αυτής της συμφωνίας δεδομένου ότι η υιοθέτηση της ε, σύμβασης θα είναι ένα σημαντικό βήμα στην δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Αντρικίνη, κυρία Κοπά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όπως πολύ σωστά είπε ο εισηγητής η περιφερειακή σύμβαση για τους πανευρωπα... Ε, ε, πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής των προϊόντων έχει σκοπό να αντικαταστήσει το εφιστάμενο δίκτυο ε, πρωτοκόλων για τους κανόνες καταγωγής να γίνει πιο ευέλικτο και πιο ξεκάθαρο η ενιαία πράξη αυτή είναι απαραίτητη γιατί κάθε φορά που πρέπει να τροποποιηθεί ένα πρωτόκολλο μεταξύ δύο χωρών εταίρων συνεπάγεται την ταυτόχρονη τροποποίηση κάθε πρωτοκόλλου που εμφανίζεται στην περιοχή αυτή. αυτή η ενιαία πράξη θα βοηθήσει πολύ και το τονίζει πάρα πολύ καλά ο εισηγητής τις χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης σε διαδικασία πολιτικών μεταρρυθμίσεων στο νότο της μεσογείου θα ήθελα να τονίσω ε, και σαν απάντηση στην κυρία Ντρικιένα και στο σχόλιο το οποίο έκανε ότι ε, είναι μια ευκαιρία με την πράξη αυτή να τονίσουμε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν σαφείς κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι ξεκάθαρα ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση στη διαδικασία τελωνιακού ελέγχου στα κράτη-μέλη της Ένωσης οι ευρωπαίοι πολίτες δικαιούνται να ξέρουν ακριβώς και με λεπτομέρεια την προέλευση κάθε προϊόντος και το ζήτημα ε, του, του ε, ισραηλινού επικισμού και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι πάρα πολύ σημαντικά. τα προϊόντα τα προερχόμενα από τα παλαιστινιακά εδάφη τα οποία είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στην επιτροπή ε, διεθνούς εμπορίου δημιουργούν λόγω του επικισμού τέτοια προβλήματα που ελπίζουμε να μπορέσουν να, σταδιακά να λυθούν. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο ο εισηγητής θέλει να σχολιάσει αυτά που άκουσε. Μπορεί, αν το επιθυμεί, διαφορετικά λίγη συζήτηση. Ο κύριος Πεγιών. Ε, απλώς να πω ότι το θέμα αυτό το πήραμε πολύ στα σοβαρά διότι ζητήσαμε την διενέργεια μιας μελέτης για αυτό το θέμα των προϊόντων που προέρχονται από τις απικίες. Είναι ένα θέμα πολύ περίπλοκο. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι γίνεται με, το, με τις τελωνιακές αρχές οι οποίες δεν μπορούν να κάνουν αυτή την επιλογή σε σχέση με τους επικισμούς. Και επειδή το θέμα είναι πολύ ευρύ ως προς την απλούστευση, προσπαθήσαμε να εξελιχθούν κάπως τα πράγματα. Το θέμα αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και θα πρέπει να μετρήσουμε την ε, περιπλοκότητά του και την ε, ανάγκη να προχωρήσουμε. Κατανοώ ότι υπάρχουν δυσχέρειες, αλλά θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε θετικά γιατί μετράει ιδιαίτερα και ο χρόνος. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Επειδή λοιπόν τελειώνουμε πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλέπαμε. Θα ήταν σκόπιμο να διακόψουμε και θα ξαναρχίσουμε στις 4 και 4 για την ακρόαση με τον κύριο Μαχμούτ Τσιμπρίλ από το ε, Διοικητικό Συμβούλιο, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου. Θα το πούμε στις 4 και 4. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Bene, cari colleghi, eh, <clears throat> credo συνάδελφοι, νομίζω ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουμε περαιτέρω, διότι έχουμε εδώ τον ε, διακεκριμένο προσκεκλημένο μας, ο οποίος ήρθε στην ώρα του. Αυτό είναι το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θα μιλήσουμε με τον δόκτωρα Μαχμούτ Τζιμπρίλ, που είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο και η συνάντηση αυτή γίνεται από κοινού με την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ. Ε, κύριε Τζιμπρίλ, θα ήταν σκόπιμο να μιλήσουμε για την παρούσα κατάσταση στη Λιβύη. Εσείς μπορείτε να μας εκφράσετε την άποψή σας όπως κρίνετε κατά τον καλύτερο τρόπο δηλαδή που κρίνεται και θα ήταν σκόπιμο να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις. Πρόσφατα μεταβήκατε στην Κίνα και θα ήθελα να μας πείτε πώς εξελίχθηκε η συνάντησή σας. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα επικαιρότητας, δηλαδή της κατάστασης στη Λιβύη όπως επικρατεί όπως έχει τώρα τελευταία. Τι προβλέπει το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο και ποιες είναι οι προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας. Πριν από την συνάντηση της Διεθνούς Ομάδας για τη Λιβύη που θα λάβει χώρα στην Ισταμπούλ την επόμενη Παρασκευή. Σας δίνω άμεσα το λόγο για να μας εκθέσετε τις απόψεις σας. Ε, ε, Ευχαριστώ. Είναι τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας να ανταλλάξω απόψεις με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Πριν από τέσσερις περίπου μήνες ήρθα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ζητήσω να ε, ε, κάνω έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας συνδράμει να σώσουμε τις ζωές των αμάχων στη Λιβύη. Σήμερα θα μπορούσα να πω ότι η κατάσταση συνεχίζεται. Η μηχανή του θανάτου εξακολουθεί να θερίζει εξακολουθεί να κάνει αυτό που έκανε για πριν από πέντε μήνες. Εμείς εξακολουθούμε να ορθώνουμε τα σώματά μας ε, προασπίζοντας τις ζωές και τα δικαιώματά μας. Η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να, προστατεύει, να προσπαθεί να προστατεύσει τις ζωές των αμάχων στη Λιβύη ενώ το καθεστώς παραμένει ε, κοφεύει σε οποιαδήποτε λογική ε, λύση ε, σε, κοφεύει σε, σε κλίση για οποιαδήποτε ειρηνική επίλυση του ζητήματος. Συνεπώς, από πολιτικής πλευράς, πιστεύω ότι αν η διεθνής κοινότητα μπορούσε να μιλήσει με μία φωνή και να συνενώσει τις ε, προσπάθειές της ε, να μιλήσει με μια φωνή και να καταδικάσει αυτές τις ε, ε, παράνομες πρακτικές, την παράνομη συμπεριφορά του καθεστώτος. Μαζί με τη, ενώ και αν παράλληλα μπορέσει να μας υποστηρίξει και στρατιωτικά, έτσι ώστε οι δικοί μας μαχητές να υπερνικήσουν τις αντίπαλες δυνάμεις, τότε θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε. Ε, χρειαζόμαστε βέβαια επίσης περισσότερη συνοχή, περισσότερη υποστήριξη, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλους τους υπέρμαχους της δημοκρατίας και της ελευθερίας στον κόσμο. Νομίζω ότι η επανάσταση της ε, Λιβύης ε, βρίσκεται σήμερα σε ένα σταυροδρόμι και οι μαχητές της ειρήνης και της δημοκρατίας πρέπει να ορθώσουν το ανάστημά τους και να μας ε, συνδράμουν με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο έτσι ώστε να ε, ε, επικρατήσει η δημοκρατία. Όταν η επανάσταση επικρατήσει στη Λιβύη δεν θα ωφεληθεί μόνο ο Λιβανέζικος λαός, ο Λιβικός λαός, συγγνώμη, θα βοηθήσει ε, να επικρατήσουν επαναστάσεις και στην ε, την Ισία και την Αίγυπτο. Ε, ταυτόχρονα αυτό θα αποτελέσει νίκη όλων, κάθε φωνής της δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή και παντού στον κόσμο. Αν η επανάσταση της Λιβύης αποτύχει, πράγμα που απευχόμεθα, αν αποτύχει να επιβάλλει μια συμμετοχική δημοκρατία, πολυφωνική δημοκρατία, μια ε, συμμετοχή στην ε, πολιτική ισότιμη για τα δύο φύλλα, αν αποτύχει η επανάσταση, τότε θα περάσουν πολλές δεκαετίες πριν ξαναεπικρατήσουν οι φωνές της δημοκρατίας ε, στην περιοχή. Συνεπώς, αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο κάτι σχετικό με τη Λιβύη, αλλά είναι η δημοκρατία στην ε, Μέση Ανατολή και στον Αραβικό κόσμο. Ε, διακυβεύονται τα συμφέροντα όλων όσοι ε, υποστηρίζουν την δημοκρατία και τις ελευθερίες στον κόσμο. Η Λιβύη είναι μια πολύ πλούσια χώρα. Έχει φυσικό πλούτο και ανθρώπινο δυναμικό. Ε, η χώρα αυτή όμως έχει στερηθεί των ευκαιριών, των δυνατοτήτων να επιλέξει το μέλλον της. Έχει στερηθεί της δυνατότητας να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά της. Ο λαός της Λιβύης ε, ε, ε, ε δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να οικοδομήσει μια χώρα με την κατάλληλη εκπαίδευση, με υποδομές, υγεία, απασχόληση για όλους, για όλους που δεν είναι παραπάνω από 6.300.000 άτομα. Και πάνω απ' όλα ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για όλους τους Λίβιους πολίτες στην ε, πολιτική διαδικασία. Ε, την ευκαιρία να ακούγεται η φωνή όλων. Συνεπώς το διακύβευμα δεν είναι μόνο λιβικό. Είναι ανθρώπινο, πανανθρώπινο παγκόσμιο. Γιατί η Επανάσταση αυτή συμβολίζει όλες τις αρχές τις οποίες ε, πιστεύουν οι δημοκρατικές δυνάμεις προσπαθούν να επικρατήσουν. Η κατάσταση στην Λιβύη σήμερα ε, είναι η Είναι αρκετά ρευστή καταρχήν γιατί υπάρχουν πολλές ε, ιδέες και ιδεολογίες αλλά και, και επιπλέον ε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη βάση για μια λύση. Ε, δύο είναι οι βασικοί άξονες μιας τέτοιας λύσης. Θα έπρεπε να είναι για να γίνει δεκτή από το λαό. Ε, η πρώτη βάση, η ο πρώτος άξονας είναι ε, η ανακοχή από την πλευρά του, της, του μηχανισμού του Κατάφη και ο δεύτερος άξονας είναι να ικανοποιηθεί η προσδοκίες του λιβικού λαού. Ο Καντάφη θα πρέπει να σταματήσει ε, τον ε, πόλεμο και να ανοίξει ανθρωπιστικούς ε, διαδρόμους, ανθρωπιστικές διόδους για να φτάσει η βοήθεια παντού. Ε, οποιαδήποτε λύση δεν ικανοποιεί αυτούς τους δύο, αυτές τις δύο προϋποθέσεις δεν θα πετύχει. Συνεπώς σας καλώ να υποστηρίξετε τον ε, λιβικό λαό στις προσπάθειές του. Να αναζητήσουμε μια πραγματική πολιτική λύση, να δοθεί ένα τέλος στην αιματοχυσία που ξεκίνησε και συνεχίζεται από τον ε, δολοφονικό μηχανισμό του καθεστώτος του Καντάφη και να δώσουμε μια ευκαιρία στη λογική να επικρατήσει. Να ικανοποιηθούν οι λογικές απαιτήσεις ε, και ε, οι θεμητές απαιτήσει του λιβικού λαού. Σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, είναι λυπηρό το γεγονό ότι η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. <clears throat> Πάνω από 450.000 Λίβοι αυτή τη στιγμή ζουν στην Τινησία. Ε, έφυγαν από την, εγκατέλειψαν την Τρίπολη, ε, την, ε, τα δυτικά όρη, τη Μιστράτα και ζουν εξόριστοι στην Τινησία ε, όπου στερούνται βασικών αγαθών όπως ε, φάρμακα τροφής, νερού, στέγης, ε, ρούχων κλπ. Οι 140 δισεκατομμύρια δολάρια είναι τα κεφάλαια της χώρας που έχουν παγώσει στο εξωτερικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν μια τόσο πλούσια χώρα έχει τόσους ανθρώπους σε ένδια και έρχεται και το Ραμαζάνι. Η κατανάλωση αυξάνεται κατά 80% στη Λιβύη τέτοιες μέρες ε, όπως και σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες ε, και ε, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι μας έχουν να πληρωθούν εδώ και δύο μήνες δεν έχουν ε, με τι να θρέψουν τις οικογένειές τους αν δεν ικανοποιηθούν αυτές οι οικονομικές ανάγκες το συντομότερο δυνατό ενδεχομένως θα ζήσουμε άλλη μια τραγωδία που θα προσθεθεί στις τραγωδίες που, έχουν προκαλέσει, που έχει προκαλέσει το καθεστώς του Καντάφη. Αυτή όμως η τραγωδία θα έχει ε, προκληθεί από εμά τους ίδιους και όχι από τον Καντάφη. Τώρα αναφορικά με τα οικονομικά ζητήματα. Ε, για να λυθούν οι για να αντιμετωπιστούν η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αναλογιστεί ότι η πρώτη προτεραιότητα για όλους είναι οι ανθρώπινες ζωές. Δεν έχει νόημα να ξοδεύουμε εκατομμύρια εκατομμυρίων δολαρίων μέσω διαφόρων διόδων για να προστατεύουμε τις ανθρώπινες ζωές από τους βομβαρδισμούς του καθεστώτος του Καντάφη και ταυτόχρονα να τους αφήνουμε να πεθαίνουν από πείνα ή από έλλειψη φαρμάκων ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης την κατάλληλη στιγμή. Έχουμε εκατοντάδες παραδείγματα ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους επειδή δεν τους δόθηκε το κατάλληλο φάρμακο την κατάλληλη στιγμή. I think about the human... Οπότε μιλάμε για την ανθρώπινη, την πολιτική, τη στρατιωτική διάσταση. Αν τις προσθέσουμε όλες αυτές, μιλούμε για μια τραγωδία την οποία υφίσταται ο λιβικός λαός εδώ και σχεδόν πέντε μήνες. Οπότε και πάλι κάνω έκκληση στην ανθρώπινη συνείδησή σας και στις πολιτικές σας αρχές που ε, είναι αρχές δημοκρατίας. Να σταθείτε δίπλα μας και να συνεχίσετε να μας υποστηρίζετε έτσι ώστε ο λιβικός λαός να επικρατήσει και να ανακτήσει την χώρα του. Σύμφωνα με τις ε, θεμητές ε, απαιτήσει ε, που προβάλλει. Για μία ακόμα φορά σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το, την ευκαιρία να σας ενημερώσω για την κατάσταση. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Τζιμπρίλ. Επτά είναι οι ομιλητές που ζήτησαν το λόγο. Θα τους δω με τη σειρά που υπέβαλαν την, το αίτημα και όχι με βάση τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Βανόρντεν να μην υπερβεί παρακαλώ τα τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Τζιμπρίλ και πάλι. Κύριε Τζιμπρίλ, μπορείτε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο. Πώς λειτουργεί, ποιους περιλαμβάνει, κατά πόσο εκπροσωπεί και ποιον εκπροσωπεί. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με άλλους Λίβιους οι οποίοι είναι εξόριστοι για πολλά χρόνια, κατά πόσο υπάρχει δηλαδή μια συμπαγής αντιπολίτευση ως προς τους εξόριστους. Την ε, Τρίτη είδαμε ότι οι απεσταλμένοι του Γκαντάφη ήρθαν σε επαφή με εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και ανέφεραν ότι θέλουν να εγκαταλείψει την εξουσία. Είναι αξιόπιστες αυτές οι πηγές. Αυτή τη στιγμή τρία αραβικά κράτη συμμετέχουν στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Άρα το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι περισσότερο για να ε, επηρεάσετε και άλλα μέλη του Αραβικού Συνδέσμου για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή στη Λιβύη. Και ποιο είναι το μήνυμά σας προς χώρες όπως η Πολωνία και η Γερμανία που έχουν ε, στρατιωτικό εξοπλισμό αλλά δεν συνεισφέρουν στην, στις επιχειρήσεις αυτές. Τι θα γίνει με την λιποταξία εκείνων οι οποίοι ακόμα υποστηρίζουν τον Καντάφη. Υπάρχουν υψηλοί αξιωματούχοι που δεν είναι στο στενό του κύκλο, αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο θα υπήρχε μία περίπτωση χορήγησης αμνηστίας έτσι ώστε να δούμε πώ θα κινηθούν ω προ ενδεχόμενη λιποταξία. Για δύο λεπτά μιλήστε κύριε Βανόρντεν, εξαιρετικά. Δεσσαρνές. Κυρία Δεσσαρνέ, ευχαριστώ ε, πρόεδρε. Όλοι ε, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχεί που σας ξαναβρίσκουμε εδώ σήμερα και ακούμε την έκκλησή σα για την υποστήριξη ε, της Ενωμένης ΕΕ Ευρώπης και της διεθνούς κοινότητας ενωμένη να υποστηρίξουμε τη Λιβική Επανάσταση. Όλοι ελπίζουμε και ευχόμαστε να πετύχει. Είναι σημαντικό για όλους τους δημοκράτες όπου και αν βρίσκονται, στη Λιβύη, στην Ευρώπη ή αλλού στον κόσμο. Έχουμε λοιπόν την ίδια αποφασιστικότητα. Θα ήθελα να σας κάνω τις εξής δύο ερωτήσεις. Η γαλλική διπλωματία εχθές δήλωσε, αν δεν απατώμε, ότι μια πολιτική λύση άρχισε σιγά σιγά να σχηματοποιείται. Αυτή είναι η ακριβής διατύπωση. Θα σας παρακαλούσα να μας πείτε εσείς τι φρονείτε. αυτό ξέρω ποιες είναι οι απαιτήσει σας για την ενδεχόμενη έναρξη πολιτικών διαπραγματεύσεων και το κατανοώ. Πάντως εσείς βλέπετε κανένα περιθώριο λιγμών και αν και η δεύτερη ερώτηση μου αφορά κάτι ε, διαφορετικό. Ε, την ΑΚΜΗ, την ε, Αλκάιτα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ. Ακούμε ότι η ΑΚΜΗ έχει στα χέρια της βαρύ οπλισμό από το στρατό του Γκαντάφη και συγκεκριμένα πυράβλους. Και τους περνάει και η ιδέα ενδεχομένως να προσπαθήσουν να αποσταθεροποιήσουν ή να εκμεταλλευτούν την κατάσταση σήμερα τη μη σταθερή στη Λιβύη και καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι αυτή η υπόθεση και θα ήθελα να μας πείτε και τη γνώμη σας και την ανάλυση σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τρία λεπτά κυρία Μπράντνε. στα αγγλικά. Ε, σας ε, καλωσορίζω και ε, σας ε, ευχαριστώ και εγώ. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι αυτό που ρώτησε η κυρία Δεσσαρνές ε, για την εκεχηρία κατάπαυση του πυρός. Ξέρω ότι έχετε βάλει ως όρο να αποχωρήσει ο Καντάφη, αλλά υπάρχει κανένα περιθώριο εκεί, ο ελιγμών. Και για σας ποια είναι τα ενδεχόμενα οι επιλογές. Λέτε ότι πιέζουν όλο και περισσότερο τα οικονομικά ζητήματα. Έρχεται και τώρα Μαζάνη. Και τι θα γίνει με τους βομβαρδισμούς, θα συνεχιστούν, θα σταματήσουν, θα πρέπει να συνεχιστούν. Και τι θα γίνει με την ε, ε, ζώνη αεροποκλεισμού. Και πώς θα πρέπει ρεαλιστικά τώρα να φανταστούμε μια πολιτική διαδικασία για την κατάπαυση του πυρός. Τι ζητάτε να μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε καμιά διαδικασία παρακολούθησης, ελέγχου, να είναι ενεργός ε, πρωταγωνιστής βεβαίω υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, να παίξει κάποιο ρόλο θέλετε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ορισμένα κράτη-μέλη. Βλέπε Γαλλία, Γερμανία θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Ποιοι είναι οι όροι σας και θα μπορούσε να σας βοηθήσει η Ένωση, αλλά με ποιο τρόπο. Και η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με το εξή. Μιλήσατε για τη μετάβαση στη δημοκρατία και γνωρίζω ότι ε, πονείτε ή επεξεργάζεστε και ένα σύνταγμα αυτό τον καιρό. Πόσο έχει προχωρήσει, ε, μέχρι πού έχετε συμφωνήσει για μελλοντικό σύνταγμα της χώρας. Πώς πηγαίνουν εκεί οι εργασίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για να υπάρχει περισσότερος χώρος για απαντήσεις, θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον πρόεδρο Τζιμπρίλ και θα συνεχίσουμε μία συζήτηση με τρεις παρεμβάσεις αναφορά και μετά απάντηση. Let me start uh, uh, Ως προς το πρώτο γύρο ερωτήσεων και ως προς την ε, σύνθεση του Εθνικού Μεταβατικού μετόπου, όταν, Συμβουλίου, συγγνώμη, όταν η Επανάσταση άρχισε τις ε, πρώτες δέκα μέρες μετά τη σύσταση του Μεταβατικού Συμβουλίου είχαμε μόνο δέκα μέλη. Οκτώ μέλη. Και συνέχεια έγιναν 31. Αυτή τη στιγμή έχουμε 49 μέλη που εκπροσωπούν ολόκληρη την ε, περιοχή της Λιβύης εκτός από τέσσερις πόλεις τις οποίες καλέσαμε, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει στείλει έναν εκπρόσωπο. Υπάρχουν διαφορές σε αυτά τα τοπικά συμβούλια για το ποιος θα πρέπει να εκπροσωπήσει τις πόλεις αυτές στο Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο. Κατά τα άλλα έχουμε 49 ε, μέλη που εκπροσωπούν ολόκληρο τον, ε, ολόκληρη την επικράτεια της Λιβύης. Το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο υπέβαλε έναν οδικό χάρτη κατά τη δεύτερη ομάδα επαφών στην Τόχα όπου προβλέπεται μια δημοκρατική κοινότητα με βάση το δίκαιο, το σύνταγμα όπου όλοι θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής χωρίς κανέναν αποκλεισμό, χωρίς τον αποκλεισμό καμίας πολιτικής δύναμης και σκιαγραφίσαμε αυτό τον οδικό χάρτη μέσα σε τρεις-τέσσερις σελίδες που δόθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στα μέλη της διεθνούς κοινότητας που έλαβαν, που συμμετείχαν σε αυτή την εκστρατεία υπέρ της Λιβύης ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκδώσει και ένα άλλο έγγραφο για την διαδικασία σταθεροποίησης όταν πέσει αυτό το καθεστώς, όπου μιλάμε για εθνική συμφιλίωση, για το πώς μπορούν να οικοδομηθούν μέτρα εμπιστοσύνης, πώς να ισχύσει ένα κράτος δικαίου, μια σωστή διάρθρωση και εκπροσώπηση ολόκληρης της επικράτητας και των πολιτικών κομμάτων που θα διανεμηθεί στην Ισταμπούλ κατά την προσεχή μας συνάντηση. Και τώρα προς τα πού κινούμαστε. Μάλλον αυτό το έγγραφο θα δείτε προς τα ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Τώρα, ως προς το γεγονός ότι ο Καντάφη λέει ότι προτίθεται να εγκαταλείψει την εξουσία, όταν το δω θα το πιστέψω. Εάν υλοποιηθεί ε, κάτι τέτοιο, τότε θα το υποστηρίξουμε κατά 100% γιατί έτσι δεν θα υπάρξει περαιτέρω αιματοχυσία, η διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης θα είναι πιο σύντομη και θα μπορέσουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας πραγματικά, στα πραγματικά ζητήματα. Στην ανοικοδόμηση της Λιβύης χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή του αραβικού κόσμου. Όπως ξέρετε, στην ομάδα επαφών υπάρχουν έξι αραβικές χώρες, συμμετέχουν έξι αραβικές χώρες δύο εκ των οποίων συμμετέχουν ενεργά στην εκστρατεία προστασίας των ανθρωπίνων, της ανθρώπινης ζωής. Πρόκειται για, για το Κατάρ και τα Εμμυράτα. Θα ήθελα να σας πω ότι η απόφαση ψηφίσματος 1973 του Συμβουλίου Ασφαλείας για την No Flying Zone Ε, οδήγησε και στην αντίδραση του Αραβικού Συνδέσμου που ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη, είχε ζητήσει από τα Ηνωμένα Έθνη να επιβάλλουν μία ζώνη απαγόρευσης ε, πτήσεων. Άρα η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν όμως τρεις ή τέσσερις χώρες που λάμπουν δια της απουσίας τους. Οι περισσότερες όμως αραβικές χώρες υποστηρίζουν τη Λιβύη και τον λαό της Λιβύης. Τώρα, ως προς την Πολωνία και τη Γερμανία, το θέμα είναι καθαρά εθνικό. Θέμα εθνικής κυριαρχίας και απόφασης. Η κάθε χώρα αποφασίζει όπως ε, κρίνει καλύτερα για να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα. Ήμουν στη Γερμανία δέκα μέρες πριν και ο Υπουργός Εξωτερικών ερωτήθη κατά πόσο ε, έχει μετανιώσει γιατί δεν υποστήριξε το ψήφισμα 1973 και είπε το γεγονός ότι δεν υποστηρίζουμε το ψήφισμα δεν σημαίνει ότι είμαστε ουδέτεροι σε αυτή την εκστρατεία ή στη σύραξη γενικότερα της Λιβύης. Ο καθένας μπορεί να, να υποστηρίξει αυτά που θέλει στα, στα κατάλληλα φόρα εκεί όπου κρίνει δηλαδή. Δηλαδή επαφείται σε κάθε χώρα να αντιδράσει όπως και όπου θέλει. Το θέμα της λιποταξίας είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τον κύκλο του Καντάφη. Εμείς αποστήλαμε, ε, ήρθαμε μάλλον σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους και μιλήσαμε για μια κατάσταση αμνηστίας, μια κατάσταση συγχώρεσης και συμφιλίωσης. Είπαμε δηλαδή ότι θα χορηγηθεί αμνηστία εκτός από εκείνους ε, τα χέρια των οποίων έχουν βαφεί με αίμα ή που αποδείχτηκε ότι είχαν συμμετάσχει σε γενικότερη διαφθορά, σε βασανιστήρια. Διαφορετικά είμαστε ανοιχτοί και δεχόμαστε τους πάντες, τα, τα παιδιά μας, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες, για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Λιβύης. Λέμε ότι θα ισχύσει ένα κράτος δικαίου και γνωρίζουμε βεβαίως ότι μερικοί Αμερική προέβαλαν βασανιστήρια, τα υποστήριξαν. Βεβαίως αυτό θα το κρίνουν ε, τα δικαστήρια, θα αποφανθούν τα δικαστήρια και όχι εμείς. Δεν είναι θέμα του Μεταβατικού Συμβουλίου. Ως προς τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλικής Κυβέρνησης, ε, πρόκειται για μια πολιτική επίλυση του ζητήματος εν εξελίξη. Βεβαίως ε, ύπτανται, περιύπτανται πολλές ιδέες γύρω από τις ομάδες επαφών. Ελπίζω να φτάσουμε σε μια πραγματική διεθνή πρωτοβουλία όπου η διεθνής κοινότητα θα εκφράζεται με μία φωνή και με μία προοπτική για να επιληθεί αυτό το θέμα της ανθρώπινης τραγωδίας που ζει η Λιβύη. Υπήρχαν και προγενέστερες ε, πρωτοβουλίες, αλλά ήταν θνησιγενείς, είτε ήταν, προέρχονταν από τον αφρικανικό χώρο, είτε όχι. Γιατί πολλές φορές λείπουν ορισμένα στοιχεία της εξίσωσης. Ελπίζω στην Ισταμπούλ να υπάρξει μία πραγματική εκπροσώπηση της διεθνούς κοινότητας η οποία να μιλήσει με μία φωνή. Εάν λοιπόν ε, συμπέσουν αυτά τα δύο στοιχεία του ψηφίσματος 1973, δηλαδή άμεση κατάπαυση του πυρός και δυνατότητα διεξαγωγής εκλογών έτσι ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να ζήσουν σε μια ελεύθερη Λιβύη, τότε νομίζω ότι όλοι θα συνέδραμαν προς αυτή την κατεύθυνση σε σχέση με τη δράση της Αλκάιντα στο Μαγκρέμπ, Νομίζω ότι ορισμένα τα, ότι η παράνομη ε, διακίνηση όπλων γίνεται μέσω του Αλγερίου. Και νομίζω ότι ε, έφυγαν από στρατιωτικούς καταβλισμούς του Καντάφη. Αυτό σημαίνει ότι ε, αν δεν ε, υφίσταται πια ο Καντάφη ως οντότητα, τότε η Αλκάιντα θα μπορέσει να δράσει ανενόχλητα στις χώρες του Μαγκρέμπ και να προωθήσει την έννοια, το σκεπτικό ότι θα πρέπει ο Καντάφη να παραμείνει στην εξουσία. Αυτή είναι η συλλογιστική που προωθείται. Αυτό όμως, αυτό το σκεπτικό απορρίφθηκε, ήταν κάτι το προκατασκευασμένο και γνωρίζουμε ότι αυτά τα όπλα τα διακίνησαν οι ίδιες οι δυνάμεις του Καντάφη για να βοηθήσουν στην επέκταση της τρομοκρατίας. Άρα η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ορθώσει το ανάστημά της κατά αυτής της ανεύθυνης συμπεριφοράς. Ως προς την κατάπαυση του πυρός, που είναι απαράβατος όρος για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις και πώς θα πρέπει να οριστεί, πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάπαυση του πυρός. Νομίζω ότι αυτό ισχύει όταν μιλάμε για δύο αντίπαλους στρατούς. Αυτή τη στιγμή όμως Μιλάμε για τον ε, ε, θανατηφόρο μηχανισμό του Καντάφη, για το ότι θα πρέπει να σταματήσει να δρά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στη Βενγάζη και αλλού σε άλλα μέρη της επικράτειας άρχισαν ειρηνικές διαδηλώσεις και προσέφυγε στη βία αποκλειστικά η κυβέρνηση, αυτό το καθεστώς, χρησιμοποίησε τα όπλα για να αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές. Δεν μιλούσαμε δηλαδή για εμπόλεμο αγώνα. Δεν ήταν αυτή η επιλογή μας. Ποτέ δεν υπήρξε. Εάν είχαμε εμείς την επιλογή στα χέρια μας, τότε θα προσφεύγαμε πάντα σε ειρηνικές διαδηλώσεις και τίποτα άλλο. Δεν θα προσφεύγαμε ποτέ στα όπλα. Εάν τώρα κατάπαυση του πυρός σημαίνει λήξη των εχθροπραξιών και μη συμμετοχή του ΝΑΤΟ πλέον, αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουν τα Ηνωμένα Έθνη, η δυνάμη του ψηφίσματος 1973, αν δηλαδή πληρούνται οι στόχοι ή όχι. Αλλά εμείς ως Λίβοι θεωρούμε Καταρχήν ότι θα πρέπει να μην προσφύγουμε στη βία, έχουμε θεμητά αιτήματα, προβάλλουμε ειρηνικές διαδηλώσεις και θα τα προβάλλουμε πάντα αυτά τα αιτήματα, ακόμα και αν χυθεί η τελευταία ρανίδα αίματος, έτσι ώστε να ζήσουμε σε μια ελεύθερη και δημοκρατική χώρα. Άρα Θεωρούμε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο για να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση και για να μπορέσουμε να ελευθερώσουμε και τις πόλεις τις οποίες, στις οποίες έχει βάλει ο Καντάφη αυτή τη στιγμή και οι οποίες πολιορκούνται από τον Καντάφη. Όμως θα πρέπει να καλύψουμε όλα τα μέρη της εξίσωσης, δηλαδή ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε μια δημοκρατική διαδικασία και αυτό προαπαιτεί την αποχώρηση του Καντάφη και της οικογένειάς του γιατί ε, έχει χάσει κάθε, κάθε ψυχείο ε, νομιμότητας πια αυτή η κυβέρνηση. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα μπορούσε να ε, εποπτεύσει την κατάπαυση του πυρός. Αυτό έγκυται στις διαπραγματεύσεις. Υπάρχει ε, ένα ευρύτερο φάσμα συμμετοχής της ε, διεθνούς κοινότητας και αυτό που έχει σημασία είναι να δεχτούμε αυτό το ευρύ φάσμα, δηλαδή είναι καλύτερα να έχουμε περισσότερες οργανώσεις παρά μία. Και βεβαίως χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από το να είχαμε την υποστήριξη μίας ή δύο χωρών. Νομίζω ότι απάντησα καταρχήν στα ερωτήματά σας. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ο κύριος Χατζηγεωργίου. Τρία λεπτά, μην τα υπερβείτε, παρακαλώ. Καταρχήν να καλωσορίσω τον κύριο Τζεμπρίλ και να του πω ότι η εισαγωγή του αλλά και οι απαντήσεις που έχει δώσει τώρα μπορεί να μην δίνουν τελικές απαντήσεις αλλά δείχνουν ότι υπάρχει τουλάχιστον μια φωνή σύνεσης και λογικής ε, γύρω από αυτό το ζήτημα. Θέλω να πω ακόμα ότι εμείς εδώ δεν είμαστε για να δώσουμε απαντήσεις, μπορεί να μην τις έχουμε και μπορεί να μην τις έχει τελικά ούτε ο κύριος Τσεπριλ. Όμως είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ανοιχτά και ειλικρινά ε, θέλω να βάλω λοιπόν μερικές σκέψεις και να δω την αντίδραση του κυρίου Κεπρίλ. Υπάρχει δυνατότητα από την παρέμβαση των δυνάμεων που έχουν παρέμβει στη Λιβύη να δώσουν τελικά το δημοκρατικό πολέτευμα που αναζητούν οι Λίβοι. Έχω την εντύπωση και θα το πω ότι δεν εμφορούνται, δεν είναι φανερό ότι εμφορούνται οι δυνάμεις που επενέβησαν σήμερα στη Λιβύη από την πίστη τους στη δημοκρατία. Εάν ήταν έτσι, θα είχαν με κάποιο τρόπο δείξει αυτό το ενδιαφέρον τους για τη δημοκρατία στη Λιβύη πριν ξεκινήσουν οποιασδήποτε αντιδράσεις μέσα στην ίδια τη Λιβύη. Αντίθετα, έχουμε την κορύφωση ενός πολιτικού αμοραλισμού όπου ετοιμάτω ο κύριος Γκατάφη μέχρι την προτεραία ε, των εξεγέρσεων και την συμφωνία μεταξύ Αγγλίας και του καθεστώτος του κυρίου Κατάφη για την ε, αποφυλάκηση ε, του συγκεκριμένου βομβιστή που ήταν στις φυλακές της Αγγλίας. Άρα εσείς κατά την άποψή μου καλά κάνετε να έχετε έγνοια για το πώς θα έρθει η δημοκρατία και θα φύγει ο Κατάφη. Αλλά πιστέψτε με την ίδια ώρα πρέπει να έχετε και μια αμφιβολία για το υγιές του ενδιαφέροντος που υπάρχει. Εγώ δεν πιστεύω στο ότι δεν δικαιούται κανείς να παρέμβει σε ένα γειτονικό κράτος. Δεν μπορεί να γίνονται δολοφονίες στο διπλανό σου σπίτι και εσύ να σιωπάς και να λες υπάρχει δικαίωμα σε αυτόν τον διπλανό χώρο να κάνουν ό,τι θέλουν. Όμως η παρέμβαση πρέπει να είναι τέτοια η οποία να φέρνει το αποτέλεσμα που θέλεις. Εδώ οι νεκροί αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Δεν μειώνεται το αίμα. Και έχουμε μια πρόσθεση ενός προβλήματος μετά από το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Πρέπει να στείλετε πιο καθαρό αυτό το μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναζητήσετε άλλου τύπου παρέμβαση και βοήθεια. Ευχαριστώ για τρία λεπτά, ε, κύριε Σκόβατσεφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Δόκτωρ Τζιμπρίλ, που ήρθατε ενώπιον μα σήμερα. Επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση που μας κάνατε για την κατάσταση. Είπατε ότι οι περισσότερες Αραβικέ χώρε υποστηρίζουν τα θεμητά αιτήματα ε, του λιβικού λαού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μα, Ποια είναι η τελευταία εξέλιξη, οι τελευταίες εξελίξεις του Αραβικού Συνδέσμου και της Αφρικανικής Ένωσης ε, για την εξέβριση πολιτικής λύσης. Αυτές οι δύο οργανώσεις, οι δύο οργανισμοί αυτοί θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ε, θετικά στην εξέβριση μιας ε, λύσης για την κρίση στη Λιβύη. Το Συμβούλιο σας έχει καθόλου σχέσεις με έναν εκπρόσωπο του καθεστώτος Ρωτώ συγκεκριμένα γιατί στην αρχή της Λιβυκής Επανάστασης είδαμε πολλά στρατεύματα ε, του Καντάφη να αλλάζουν πλευρά και να πηγαίνουν την πλευρά των ανταρτών. Ε, τώρα εσείς εκτιμάτε, αναμένετε να συνεχιστεί αυτή η εικόνα και στο προσεχές μέλλον, γιατί τέτοιου είδους πληροφόρηση δεν έχουμε έτσι πρόσφατη τους τελευταίους μήνες, όσο είχαμε στην αρχή. Και εκτός από την ερώτηση του αδέλφου Βαν Όρντεν. Το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο διατηρεί επαφές με τους Λιβύους εκτός της Λιβύης, στο εξωτερικό. Και πώς βλέπετε το ρόλο, το ενδεχόμενο του Ιού του Τέος Βασιλέως ε, προς ε, μια δημοκρατική Λιβύη. Και μια τελευταία ερώτηση, μια που είμαι και βούλγαρος, δεν μπορώ να χάσω την ευκαιρία να σας ρωτήσω αν αναμένετε να δεχτείτε έτσι περισσότερες προφορίες για να μάθετε τι έγινε με τις Βουλγάρες νοσοκόμες και του Παλαιστίνιο γιατρό. Αυτή την υπόθεση θυμάστε στη Λιβύη πριν από λίγα χρόνια. Όταν τους κατηγόρησαν ότι ε, μόλυναν με AIDS τα παιδιά στη Λιβύη και θυμάστε ήταν μεγάλη πολιτική αναταραχή και πρόβλημα όχι μόνο για τη Λιβύη και τη Βουλγαρία αλλά και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε καθόλου καινούργιες προφορίες. Περιμένουμε μετά τη μετάβαση προς τη δημοκρατία να μάθουμε τίποτα καινούριο. Τι συνέβη ακριβώς τότε εκείνες τις μέρες. Και αν μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες ε, προφορίες εκ των έσω. Ευχαριστώ. κύριος για τρία λεπτά. Ευχαριστώ να σας καλωσορίσω θερμά από τους Ευρωπαίους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές και θα ήθελα να τονίσω ότι θαυμάζω το θάρρος σας διότι προσπαθήσατε να απομακρύνετε αυτό τον ψυχοπαθή τύρανο με τα παιδιά του. Ελπίζω σύντομα να αποχωρήσουν. Γιατί η Αλγερία βοηθά τον Καντάφη επιτρέφοντας την ελεύθερη διακίνηση όπλων και μισθοφόρων. Φαίνεται ότι είναι η μόνη χώρα η οποία βοηθά το καθεστώς του Τρίπολης. Ως προς το θέμα της συμμετοχής της αλ ε, έγινε λόγος για μια παραφιάδα της Αλ-Κάιντα, η οποία ελπίζουμε να εξαλειφθεί. Το γεγονός ότι ζητήθηκε καταδίκη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θεωρείται ότι ήταν ε, ένα μέτρο έτσι ώστε να ε, προωθηθεί η σύλληψη του Καντάφη σύντομα ποιος θα ε, εκενώσει τους μισθοφόρους, διότι αν δεν γίνει σύντομα τότε θα λιντσαριστούν. Επίσης οι Βέρβεροι πώς δρούν και οι Γάλλοι μπορούν να τους δώσουν οπλισμό. Ποιος θα χρηματοδοτήσει την Αφρικανική ε, ε, Ένωση μέσα στα πλαίσια της, μετά τον Καντάφη εποχής. Ευχαριστούμε κύριε Τάνουκ. Ο πρόεδρος Τζιμπρίλ έχει το λόγο. Θα ήθελα να μας μιλήσει το πολύ για 9 λεπτά. Να μην υπερβεί τα 9 λεπτά. Γιατί όχι 8 ή 10. Γιατί τόσο έδωσε και στους ομιλητές. Τρεις ομιλητές από τρία λεπτά. Ωραία. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος λοιπόν. για τις ε, χώρες της διεθνούς κοινότητας που ε, επενέβησαν στην Λιβύη κατά του ψηφίσματος 1973 κανένας ε, δεν λέει ότι ήρθαν για να εδραιώσουν τη δημοκρατία. Το ψήφισμα λέει ότι ήρθαν για να σώσουν τις ζωές των αμάχων βομβαρδισμοί ξεκίνησαν από τις 17 Φεβρουαρίου και η παρέμβαση, η επέμβαση έγινε ένα μήνα μετά. Ένα μήνα και δύο μέρες μετά, στις 19 Μαρτίου ξεκίνησε για να σωθούν οι ζωές των αμάχων. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτές οι χώρες έρχονται για να σώσουν τη δημοκρατία. Πολύ απλά, διότι η δημοκρατία θα πρέπει να ανθίσει από μέσα. Δεν είναι αγαθό εισαγωγής, εισαγόμενο αγαθό αν η δημοκρατία δεν είναι κουλτούρα, δεν είναι νοοτροπία στα μυαλά και στις καρδιές των ανθρώπων, ε, ε, είναι θνησιγενής. Ε, αν εμείς μέσα μας δεν έχουμε αυτό που χρειάζεται να είναι κανείς δημοκράτης, η δημοκρατική θεσμή, εκλογή και όλα τα υπόλοιπα είναι ανεπαρκή. Συνεπώς, συμφωνώ μαζί σας ότι αυτή η επέμβαση δεν γίνεται για να ε, επιβληθεί η δημοκρατία. κανένα δεν το ισχυρίζεται αυτό. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι μετά το 2002 υφίσταται το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Η διεθνής κοινότητα λοιπόν δεν μπορεί ε, να ε, εθελοτυφλεί μπροστά σε τέτοιου είδους τραγωδίες ανθρωπιστικής φύσεως ε, οι οποίες ε, γίνονται όλο και πιο ε, ορατές μέσω του ίντερνετ και των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας. Αν καθόμασταν στο περιθώριο και δεν κάναμε κάτι για τέτοιου ανθρωπιστικέ τραγωδίε, θα αντιφάσκαμε τον εαυτό μα. Συνεπώ, ακόμα και οι χώρε οι οποίε δεν παίρνουν μέρο στρατιωτικά ε, στι επιχειρήσει αυτέ κάνουν το καθήκον του με άλλο τρόπο. Γιατί είναι μια τραγωδία η οποία θα πρέπει να σταματήσει. Τώρα, η Αφρικανική Ένωση. Ε, η Αφρικανική Ένωση είχε υποβάλει ένα οδικό χάρτη ε, που όμως ε, συνοψίζεται σε μια έκκληση για κατάβαση του πυρός και μια επίλυση του προβλήματος μέσω διαπραγματεύσεων. Η πρωτοβουλία αυτή δεν θέτει όμως συγκεκριμένους στόχους για τις διαπραγματεύσεις. Δεν καλεί να σε αλλαγή του καθεστώτος, αλλά σε αναμόρφωση του βελτίωση του καθεστώτος. Γι' αυτό το λόγο δεν συζητήθηκε καν από το λαό μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το ε, αν περιμένω ε, καινούριες αποστασίες. Ναι, ναι, όλο και περισσότερες. Ε, ήδη ε, έχουμε ε, τέτοιου περιπτώσεις ε, και σε ψηλοβαθμούς αλλά και σε μεσαίους βαθμούς του στρατέματος του Καντάφη. Ορισμένες τέτοιου είδους περιπτώσεις ήταν δάκτυλοι του καθεστώτος που θέλησαν να στείλουν πράκτορες τους στις δικές μας τάξεις κανένας δεν ε, εξαιρείται, ούτε αυτοί ε, που προέρχονται από το καθεστώς του Καντάφη, ε, γιατί αν τους εξαιρούσαμε θα ήταν σαν να κάναμε ό,τι κάνει ο Καντάφη. Σε ό,τι αφορά τις νοσοκόμες από την Βουλγαρία, αν επιθυμούμε την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου μετά από όλη αυτήν την ιστορία, είναι προφανές ότι οποιαδήποτε αδικία έχει διαπραχθεί ε, θα διορθωθεί ε, ξανανοίγοντας το φάκελο. Νομίζω ότι αυτό είναι δικαίωμα όλων. Ε, νομίζω ότι όλα θα πρέπει, όλες οι αδικίες που έχουν διαπραχθεί θα πρέπει να διαρευνηθούν. Γιατί η Αλγερία βοηθάει τον Καντάφη. Καταρχήν, ελπίζω ότι η, η Αλγερνοί αδελφοί μας, και δεν μιλώ για την κυβέρνηση, ε, θα ακούσουν την φωνή της λογικής και θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι την ιστορία τη γράφουν οι λαοί πάντοτε ε, και εμείς υποστηρίξαμε τη δεκαετία του 50 την επανάσταση των Αλγερινών τον αγώνα τους. Τους υποστηρίξαμε οικονομικά, λάβαμε μέρος στην επανάστασή τους δίπλα τους, ε, χύσαμε το αίμα μας πολεμώντας ε, την απεικιοκρατία. Συνεπώς δεν αξίζουμε αυτή την ε, συμπεριφορά πλευράς του αλγερνού λαού. Τώρα γιατί έχουν το, το, τους ε, λόγους τους. Ίσως η δομή της χώρας, ε, οι Βερβέροι του Νότου ε, φοβούνται ότι η επανάσταση αυτή θα περάσει τα ε, σύνορα και θα φτάσει μέχρι το Μαρόκο. Στο Μαρόκο από την άλλη μεριά γίνονται, γίνεται ε, γίνονται προσπάθειες να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Ε, η Τινησία έχει ε, ήδη κάνει την επαναστασή της, η το ίδιο. Η μόνη χώρα η οποία δεν έχει κάνει τίποτα είναι η Αλγερία. Ίσως λοιπόν η επιτυχία του, της Λιβικής Επανάστασης μπορεί να, ξεσπάσει, να επεκταθεί και εκεί. ο Καντάφη είχε την ευκαιρία από την άλλη μεριά να κάνει τις επιλογές του τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Συνεπώς ακόμα και με την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δεν ξέρω αν στριμώχνεται στην γωνία ε, και πάλι έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό που πρέπει. Την απόφαση θα την πάρει ο ίδιος όμως, όχι οποιοδήποτε δικαστήριο. Ο Καντάφη έχει το, τη δυνατότητα στα χέρια του να σταματήσει από την αιματοχυσία αμέσως Ποιο θα χρηματοδοτήσει Τούσε την Αφρικανική Ένωση μετά τον Καντάφη, στη μετά Καντάφη εποχή. Νομίζω ότι αυτή η οργάνωση που δημιουργήθηκε το 1963, πολύ πριν έρθει ο, στην εξουσία ο το 1969, ε, μπόρεσε να λειτουργήσει και πριν τον Καντάφη και θα μπορέσει να λειτουργήσει και μετά τον Καντάφη. αν η χρηματοδότηση μιας οργάνωσης εξαρτάται από έναν μόνο άνθρωπο, ε, τότε η οργάνωση αυτή πραγματικά ε, έχει πολλούς μπελάδες μπροστά της. Ευχαριστώ κύριε Τζιμπρίλ. Ε, δεν υπερβήκατε τα 9 λεπτά. Αρκεστήκατε και σε επτά για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις έγιναν τώρα, οι οποίες αφορούν τη φάση της μετάβασης εγώ θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις με μια απότερη πρόπτικη. Ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οικονομία και πώς τη φαντάζεστε. Κύριε Τζιπρίλ, μέχρι τώρα το πετρέλαιο ε, περνούσε από μια διαδικασία που ονομαζόταν ε, EPSA ε, κάθετος 4 που για τις ξένες εταιρείες ήταν ιδιαίτερα μειονεκτικό. Σκέφτεστε να το αλλάξετε αυτό ή ε, το έχετε ήδη αλλάξει. Γιατί κυκλοφορεί ήδη το πρώτο πετρέλαιο, ρέει από τις ε, περιοχές σας. Ε, θα ιδιωτικοποιήσετε τον τομέα της ενέργειας πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Επίσης, σας ρώτησαν για την Αφρικανική Ένωση, συνάδελφοι. Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω κάτι. Η Λιβύη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ε, στα οικονομικά της Αφρικανικής Υπήρου στο σύνολό της. Το, το Αφρικανικό Νομισματικό Ταμείο, Κεντρική Τράπεζα κτλ. Ε, θα διατηρήσει αυτό το ρόλο η Λιβύη ή πώς φαντάζεστε το ρόλο σας στο μέλλον. Και αν μου επιτρέψετε και μια προσωπική ερώτηση. Εσείς μετά την ολοκλήρωση της διένεξης θα είστε διαθέσιμος για ένα νέο υπουργικό θόκο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταφ. Τρία λεπτά σας παρακαλώ. Κύριε Τζιμπρίλ, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτά που λέτε δεν ακούγονται πάρα πολύ αισιόδοξα σχετικά με το ενδεχόμενο και την προοπτική μιας ε, ε, ε, διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων. Εκτιμώ πάρα πολύ τις καλές σας και φιλελληνικές προθέσεις, αλλά μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι έτσι πάρα πολύ ομά και με ευθύ τρόπο. Ποια είναι τα επόμενα στρατιωτικά βήματα που νομίζετε ότι είναι απαραίτητα για να ανατραπεί το καθεστώς Καντάφη ή μάλλον για να το πω με άλλα λόγια εσείς τι ζητάτε από το ΝΑΤΟ και μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση, ίσως και πιο εύκολη. Οι πηγές χρηματοδότησης του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου Ποιες είναι, μέχρι τώρα είχατε πρόσβαση στα διεθνή στοιχεία ενεργητικού της χώρας που έχουν παγώσει. Περιοριουσία εννοώ της οικογένειας Καντάφη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ κύριε Νταφ. Η κυρία Φλότρ, παρακαλώ, για τρία λεπτά. Θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις που μάλλον είναι δυσάρεστες. Γιατί η πρώτη αφορά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν τεκμηριωθεί και πρόσφατα και δεν είναι πρώτη φορά από την ε, Human Rights Watch ε, ότι αφορά ε, τη δράση των εξεγερθέντων. Εσείς πώς αντιδράτε σε αυτά τα γεγονότα και σε αυτές τις εκθέσεις. Θεωρείτε ότι είναι παράπλευρες ζημίες, απώλειες της σύγκρουσης ή αναλαμβάνετε την ευθύνη σας της αρχής γιατί αγωνίζεστε για το κράτος δικαίου, την ελευθερία και τη δημοκρατία. Έχετε μηχανισμούς για να αντιμετωπίσετε θεωρήσετε ότι υπεύθυνοι και υπόλογοι αυτών των τεκμηριωμένων επαναλαμβάνων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η δεύτερη ερώτηση. Εξεπλάγει πολύ όταν είδα πόσο βιαστήκατε να, να υπογράψετε με την Ιταλία συμφωνία μετανάστευσης. Εγώ πως σας θα περίμενα μάλλον σαφή έκκληση προς ευρωπαϊκές χώρες για να βοηθήσουν το ένα εκατομμύριο προσώπων που έχουν διαφύγει από τη Λιβύη και ε, που τους έχουν υποδεχθεί στο Τσάτ, στον Ήγυρα, ε, στην Αίγυπτο, στην Τινησία από πάρα πολύ αντίξωες συνθήκες. Εσείς που υπογράψατε αυτή τη συμφωνία, είστε πρόθυμοι να τους δεχθείτε πίσω που θα σας στέλνουν στις ε, περιοχές που έχετε απελευθερώσει όπως λέτε και θα σεβαστείτε και θα εγγυηθείτε και τα δικαιώματά τους. Πώς τη βλέπετε αυτή την ευθύνη την οποία δεχθήκατε υπογράφοντα αυτή τη συμφωνία με την Ιταλία. Ευχαριστούμε την κυρία Φλότρο. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Τζιμπρίλ μέχρι τελική πτώσεως. Uh, uh, Σε ό,τι αφορά την ιδιωτικοποίηση του πετρελαίου και των πετρελαϊκών εταιριών. Αυτό είναι θέμα που θα αποφασίσει ο λιβικός λαός, δεν θα το αποφασίσω εγώ. Παρακαλώ, έχετε υπόψη ότι το Συμβούλιο μας είναι μεταβατικό σώμα. Δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις ε, ξονόματος μελλοντικών κυβερνήσεων ή μελλοντικών αποφάσεων του λιβικού λαού. Το είδος, τον τύπο της οικονομίας μας, τη ταυτότητα, τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την ανάπτυξη. Όλα αυτά θα τα αποφασίσει ο λιβικός λαός. Εμείς είμαστε ένα μεταβατικό όργανο για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ε, δεν είναι θέματα στρατηγικά που θα αποφασίζουμε εμείς, αλλά ο λιβικός λαός. Ο ρόλος της Λιβύης στα πλαίσια της Αφρικής θα ήταν και θα συνεχίσει και θα παραμείνει θέμα γεωγραφίας, ξέρετε. Δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι η Λιβύη είναι η πύλη που συνδέει την Αφρική με την Ευρώπη. Είναι στρατηγική η θέση της δεν μπορεί η Λιβύη να έχει την πολυτέλεια να μην διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αφρική. Έγινε προσωπική ερώτηση αν θα είμαι διαθέσιμος μετά τη λήξη της σύγκρουσης. Όχι. Έχω υποσχεθεί, έχω δεσμευτεί ότι δεν θα παίξω κανένα επίσημο ρόλο όταν τελειώσει αυτή η δοκιμασία και έχω δεσμευτεί στο παρελθόν επίσημα και θα το τηρήσω. Ε, σε ό,τι αφορά το θέμα το τι χρειάζεται από στρατιωτικής πλευράς για να τελειώσει αυτό το μαρτύριο ε, θα σας έλεγα πρώτα απ' όλα ότι δεν είμαι απεσιόδοξος. Στο βαθμό που υπάρχει η αποφασιστικότητα του λιβικού λαού να αγωνίζεται για τα θεμητά του αιτήματα, είμαι αισιόδοξο ότι θα γίνει. Είναι απλώ ζήτημα χρόνου. Αν θα γίνει μέσω της αντίστασης στρατιωτικής ή με πολιτικά μέσα, Πόσο χρόνο θα χρειαστεί δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι ότι ο λαός έχει πάρει τις αποφάσεις του και δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι. Θα έρθει νέα Λιβύη και σίγουρα θα γίνει αυτό. Τι θέλουμε από το ΝΑΤΟ. Εδώ θα χρησιμοποιούσα τον όρο ή την έννοια στον κοινότητα, διότι ενέχονται και άλλες χώρες σε αυτή την εκστρατεία, όπου ηγείται βεβαιω το ΝΑΤΟ, αλλά συμμετέχουν και άλλες χώρες στην εκστρατεία προστασίας ε, ε, του αμάχου πληθυσμού. Μα αν συνεχίζετε... Ε, η ε, ε, δολοφονία αυτή των πολιτών θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν ε, το ψήφισμα 1973 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν θέλουν να κάνουν εκείνοι το δικό μας πόλεμο, να δώσουν τη δική μας μάχη, αλλά να γνωρίσουν τα θεμητά μας τίματα να μας βοηθήσουν πολιτικά, ηθικά και στρατιωτικά να τα πετύχουμε με κάθε μέσο. Το ΝΑΤΟ όμως ε, έχει αναλάβει το μερίδιο που του αναλογεί και συγκεκριμένα με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε στο έδαφος ε, πολιτικά με όσα μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, όλα τα εργαλεία και τα μέσα για να φτάσουμε στο στόχο μας που είναι να θυδρήσουμε τη δημοκρατία στη Λιβύη. Οι πηγές χρηματοδότησης του Συμβουλίου δεν χρηματοδοτούμαστε εμείς. Λειτουργούμε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη οικονομική κατάσταση. Διότι πάνω από 300 εκατομμύρια ε, δινάρια έχουν ε, δαπανηθεί τους τρεις πρώτους μήνες. Για δύο μήνες δεν έχουν, ε, δεν έχουν πληρωθεί οι δημόσιοι υπάλληλοι 500 εκατομμύρια δολάρια εκτιμώνται οι ανάγκες για φάρμακα το επόμενο εξάμηνο γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από φάρμακα και από τρόφιμα, μεγάλο ε, έλλειψη. Θα ενταθεί αυτό και θα φανεί πάρα πολύ έντονα το ραμαζάνι που σας είπα ότι αυξάνεται η κατανάλωση και ρούχα χρειαζόμαστε ε, τα βασικά ε, καθημερινά. Σε, ένα, σε μήνα θα ξανανοίξουν τα σχολεία και δεν έχουμε τα μέσα τα οικονομικά ε, να ε, καλύψουμε ε, στις ελεύθερες περιοχές 1,5 εκατομμύριο μαθητές. Έχουμε διάφορες συνεισφορές από Λιβύους επιχειρηματίες, από τους Λιβύους της Διασποράς, αλλά πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη στενότητα από πλευρά οικονομική, διότι τα ε, χρήματα του, του κράτους είναι παγωμένα στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ασία, σε διεθνείς ξένες τράπεζες. Και δεν μπορούμε να ε, φτάσουμε ε, στους πόρους αυτούς για να καλύψουμε τις καθημερινές ανάγκες του λαού μας για τις παραβιάσεις αυτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μεμονωμένα περιστατικά επεισόδια που έγιναν τις πρώτες μέρες της Επανάστασης. Είναι πραγματικά, ε, γίνεται, διεξάγεται έρευνα αυτό τον καιρό για να ε, διαπιστωθούν οι πέτοι και να είστε βεβαία ότι όποιος ευθύνεται γι' αυτά θα ε, έρθει ενώπιον της δικαιοσύνης. όταν ζητούμε ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία θα πρέπει πρώτα να το εφαρμόζουμε στους εαυτούς μας. Σε ό,τι αφορά το θέμα της υπογραφής συμφωνίας με την Ιταλία, το έχετε δει εσεί αυτό το έγγραφο. Σα ρωτώ, έχετε δει εσεί τέτοια συμφωνία το κείμενο. Θα ήθελα πολύ να το δω, λέει η κυρία Φλότρ. Πολύ θα ήθελα να το δω. Ε, ε, θα ήλπιζα να το είχατε δει πριν ρωτήσετε, διότι δεν ήταν συμφωνία καταρχάς, ήταν μνημόνιο συνεννόησης, δεν ήταν καμία συμφωνία για λαθρομετανάστευση καθόλου. Ήταν ένα θέμα πώς αντιμετωπίζει τη λαθρομετανάστευση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά ούτε δεσμευτήκαμε, ούτε υποσχεθήκαμε τίποτα. Ένα μνημόνιο συνεννόηση ήταν και εμεί ω Συμβούλιο δεν έχουμε δικαίωμα να υπογράφουμε ούτε συνθήκε ούτε συμφωνίε ούτε τίποτα. Ήταν ένα μνημόνιο και τίποτα παραπάνω. Για να διευκρινίσω το ζήτημα. Bene. Eh, grazie al... Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο Τζιμπρίλ. Η συνάντηση ήταν άκρος ενδιαφέρουσα και χρήσιμη και Ευχόμαστε να ξαναβρεθούμε στο εγγύς μέλλον οπότε, οπότε η χώρα σας θα έχει ακολουθήσει την διαδικασία ειρήνευσης, θα υπάρχει ειρήνη στη Λιβύη και θα ήθελα να σε ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει ε, στις 31 Αυγούστου. Να ευχαριστήσουμε και την Κομισιόν με τις ε, διακλαδώσεις της που βρίσκεται εδώ πάντα παρούσα. <laughs>